μεζικές αρχές για θέματα πολιτικής και κάναμε και μερικά πράγματα μαζί. Υπάρχουν όμως ε, κάποια άλλα θέματα που για αυτά κυρίως περιοριζόμαστε στη θεωρία και δεν περνάμε στην πράξη. Και αυτό συμβαίνει κυρίως ε, στον τομέα της οικονομίας. Η Κίνα είναι πολιτική υπερδύναμη, είναι υπερδύναμη στην εξωτερική πολιτική, στο στρατιωτικό τομέα, στην τεχνολογία, στις επιχειρήσεις, στην οικονομία σε πάρα πολλούς τομείς. Άρα δηλαδή δεν έχει νόημα να θεωρούμε την Κίνα ως αναπτυσσόμενη χώρα. Σίγουρα η Κίνα είναι αναπτυσσόμενη χώρα ε, για διάφορους άλλους λόγους, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τη δύναμή της στην παγκόσμια οικονομία σήμερα, έχουμε κάθε λόγο ε, να περιμένουμε αμοιβαιότητα. Αυτό λοιπόν περιμένουμε από την Κίνα. Να είμαστε στρατηγικοί εταίροι που βασιζόμαστε στην αμοιβαιότητα. Κυρίως όσον αφορά τις πολιτικές για την πρόσβαση στην αγορά. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούν να ε, βελτιωθούν οι οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις με την Κίνα. Και αυτή τη στιγμή σε αυτό δουλεύουμε. Παραδείγματο χάρη προετοιμάζουμε κανόνες ε, για κρατικές ενισχύσεις ε, σχετικά ε, με την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων εκτός τρίτων κρατών. Εμείς έχουμε αυστηρούς κανόνες για το ισχύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους κανόνες για τις τρίτες χώρες. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ίσους όρους για όλους. Θεμητό ανταγωνισμό και όχι αθέμητο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κοινή μας αγορά θα είναι ανοιχτή για όλους, αλλά με με δίκαιους όρους δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αθέμητο ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Επίσης, όπως είπε προηγουμένω και ο πρόεδρος κύριος Τούσκ, θέλουμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία για τις επενδύσεις σε συμφωνία με την Κίνα μέχρι το 2020. Πολύ σημαντικό. Θα βοηθήσει ευρωπαϊκές και κινέζικες επενδύσεις να ανθίσουν. Επίσης, περιμένουμε με την Κίνα να δεχτεί τη συμφωνία γεωγραφικών ενδείξεων που μέχρι τώρα συζητιέται αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί. Αξιότιμα μέλη, όπως σας είπα, είμαστε στρατηγικοί εταίροι, ε, συνεργαζόμαστε στενά σε πάρα πολλούς τομείς τομείς της πολιτικής, αλλά κυρίως η οικονομική συνεργασία είναι ένας τομέας όπου πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις για να διατηρηθούν ίση όροι ανταγωνισμού και να μπορούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες να κάνουν στην Κίνα αυτό που οι κινέζικες εταιρείες πράττουν στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ, λέει ο Πρόεδρος. Και ε, για την τελική ομιλία, τελική παρέμβαση, ο κύριος Τούσκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις. Δεν είναι αυτό το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν από τις ε, εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ πιθανό να συναντηθούμε τον Απρίλιο για να συζητήσουμε τον Brexit και σίγουρα θα συναντηθούμε και στις 9 Μαΐου στο Σύμπιου για να συζητήσουμε την μακροπρόθεσμη ενωσιακή μας πολιτική. Θα είναι άτυπη συνάντηση, αλλά θα είναι αφιερωμένη σε πολύ κρίσιμα θέματα. Κύριε Φάραντζ, μιλήσατε με πάθος ενάντια στο δεύτερο δημοψήφισμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο δημοψήφισμα έγινε το 2016 γιατί το πρώτο έγινε το 1975 και τότε η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών είχαν αποφασίσει ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Εσείς ε, θεωρήσατε ότι θα μπορούσατε να φύγετε, θα οργανώνατε ένα δημοψήφισμα για να ακυρώσετε το προηγούμενο. Και αυτό με συνέπεια κάνετε και σήμερα. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Euh, euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας με την κοινή συζήτηση για τη δέσμη ε, μέτρων κινητικότητας. Έχουμε καταρχήν την έκθεση κυλών για τι απαιτήσει επιβολή και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Έκθεση Βαντεκάμπ για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγηση κατά τα τόρια για τα διαλύματα περίοδου ανάπαυση και εντοπισμού μέσω ταχογράφων και έκθεση ΕΡΤΟΥΚ για την προσαρμογή σε εξελίξει στον κλάδο δικών μεταφορών. Το λόγο έχει πρώτα η κυρία Κιλόνεν. Arvoisa πρόεδρε, συνάδελφοι, έχει γίνει σάγκα το θέμα αυτό. και χρειαζόμαστε μεγάλη δύναμη και επιμονή για να συνεχίσω με αυτό που άρχισε πριν από δύο χρόνια. Θέλουμε δίκαιους κανόνες στις μεταφορές. Αξιοπρεπείς, σωστές κοινωνικές συνθήκες στην αγορά. Είναι μεγάλη πρόκληση το θέμα αυτό. Έχουμε καταθέσει τροπολογίες. Ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι υπερβολικές για ένα νομοθέτημα. Χρειαζόμαστε πιο αυστηρούς κανόνες όμως. Οι συμβιβασμοί ε, δεν ε, σημαίνει ότι κάποιοι θα φεύγουν ε, με το αίσθημα του νικητή. Ε, εκείνο που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να έχουμε δίκαιους κανόνες στις, ε, στον τομέα των μεταφορών που θα επέτρεπε στους οδηγούς και τις εταιρείες ε, να εργαστούν αποδοτικά. Ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση που προηγήθηκε Υπήρξαν ισχυρισμοί ότι ε, ήταν ε, πάρα, πολύ, πάρα πολλές συμβαστικές τροπολογίες. Πάντως, ε, δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ να παίζονται παιχνίδια στην Ευρώπη σε βάρος των οδηγών. Υπάρχουν... Ε, εταιρείε εικονικές που καταστρατηγούν τους κανόνες. Εμείς από την αρχή πιστεύαμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ομαδική οδήγηση. Οι οδηγοί δικαιούνται να πηγαίνουν να επισκέπτονται τις οικογένειές τους ε, όποτε επιθυμούν, να πηγαίνουν όπου θέλουν και αυτό το ελάβαμε υπόψη μας ε, στις τροπολογίες. Ε, ε, λάβαμε υπόψη μας το δικαίωμα των οδηγών να επιστρέφουν στην ε, πατρίδα τους ή σε ένα άλλο τόπο που επιθυμούν. Επίσης, η ιδέα ήταν η ίση αμοιβή για ίση εργασία. Διότι στον τομέα των μεταφορών πρέπει να τηρούμε την αρχή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Α, θα έπρεπε αυτό να ισχύει και για την απόσπαση των εργαζομένων που υπάρχουν διαφορές στις, στην αμοιβή. Πολλοί ε, θα μιλούσαν εδώ για κοινωνική προστασία, αλλά ε, πολλές φορές αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει την ευελιξία. Επίσης δεν θέλουμε ε, φορτηγά να κυκλοφορούν στην Ευρώπη χωρίς ε, φορτίο. Ε, θα πρέπει να δώσουμε τέλος στο παράνομο, στις παράνομες ενδομεταφορές και τις άλλες παράνομες πρακτικές. Η ιδέα είναι να δημιουργήσουμε σαφή, σαφείς υποχρεώσεις και σαφείς κανόνες επιβολής του νόμου. Ε, αυτό ισχύει και για τους ηλεκτρονικούς ταχογράφους και άλλα μέτρα. Η ηλεκτρονική ταχογράφη είναι σημαντική εδώ. Ε, πετύχαμε και συμβιβαστικές λύσεις. Πολλοί εργάστηκαν για να αποφύγουν ε, να ψηφιστούν οι συμβιβαστικές τροπολογίες. Εμείς θέλουμε όμως να αποδείξουμε ότι οι οδηγοί έχουν δικαίωμα για δίκαιους κανόνες και ε, επίση ε, κανόνες για να είναι ισότιμη η όριο ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Τέσσερα λεπτά ο κύριο Βαντεκάμπ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που είπε η προραλή και θέλω να σας επιβεβαιώσω ότι η δέσμη κινητικότητας είναι ένα, μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων όπου πρόκειται για την απόσπαση, για, το καποτάζ και για ώρες οδήγησης και ανάπαυσης. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, συνειδητοποίησαμε όλοι ότι πρόκειται για ένα θέμα πολιτικά πολύ ευαίσθητο. Πρόκειται για την ουσία της ε, κοινή αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στη δική μου την παρέμβαση θέλω να αναφερθώ στους όρους, στο ωράριο οδήγησης και ανάπαυσης, να βελτιωθούν οι συνθήκες. Δεν πρόκειται τόσο πολύ για το ημερήσιο πρόγραμμα οδήγησης και ανάπαυσης. Αυτό ρυθμίστε σε ένα άλλο ε, χαρτοφυλάκιο. Πρόκειται για τις ώρες οδήγησης και ανάπαυσης τη νύχτα και το Σαββατοκύριακο. Και το σημαντικότερο ερώτημα που τίθεται είναι ο οδηγός που ακριβώς ε, θα περνάει αυτές τις ώρες. Διαπιστώσαμε ότι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλούς ευρωπαϊκούς δρόμους έχουμε παράνομη στάθμευση. Εκεί δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις υγιεινής, δεν υπάρχουν ε, κουζίνες. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα λύσουμε με την ε, έκθεσή μας και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μεγάλο βαθμό μα στηρίζει, αλλά το Δικαστήριο είπε επίσης ότι οι χρόνοι ανάπαυση δεν πρέπει να λαμβάνουν χώρα στον θάλαμο του οδηγού. Ε, εμείς ε, δεν μπορέσαμε να το απαγορεύσουμε, θελήσαμε να βρούμε μια μεταβατική λύση. Και τίθεται το εξή ερώτημα. Ο οδηγό πότε ε, θα μπορεί να επιστρέφει στο σπίτι του, γιατί δεν θέλουμε οδηγού νομάδε οι οποίοι να λείπουν εβδομάδες ολόκληρες από τα σπίτια τους. Θα πρέπει να μπορούν να επιστρέφουν στα σπίτια τους σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτό πρέπει να το εγγυάται ο νομοθέτης. Έχω κατά νου, παραδείγματος χάρη, τουλάχιστον κάθε τέσσερις εβδομάδες. Και επίσης ε, να υπάρχει χρόνος ανάπαυσης ε, για κάθε εβδομάδα σε ε, χώρους στάθμευσης με ικανοποιητική εγκατάσταση. Κάτι άλλο, η οδηγή λεωφορείων. Κυρία Πρόεδρε. Ξέρετε ότι ε, αυτά δεν είναι εμπορευματοκιβώτια. Γι' αυτό λοιπόν για τους οδηγούς λεωφορείων θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία, όχι 16 ώρες οδήγησης, όπως λένε μερικοί σοσιαλδημοκράτες. Θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την περίφημη ρύθμιση των 12 ημερών. Κυρία Πρόεδρε, ένα σημαντικό θέμα σε αυτή την έκθεση είναι η εφαρμογή. Η κυρία Κιλόνεν το έθιξε ήδη το θέμα και εμείς όλοι επιθυμούμε προτιμούμε την 1η Ιανουαρίου του 2024 να υπάρχει ο περίφημος ευφύης ταχογράφος δεύτερης γενιάς. Ισχύει το εξής και οι εικονικές εταιρείε και αυτές ε, πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τελειώντας, θέλω να πω κάτι για το καμποτάζ και για την απόσπαση. Πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να μην έχουμε πολύ αυστηρούς νόμους. Γιατί με αυστηρούς νόμους παρεμποδίζεται, παρακολύεται η εύρυθμη λειτουργία της κοινή αγοράς. Αυτή τη στιγμή λείπουν πάρα πολλοί οδηγοί. Έχουμε ε, λιγότερους, λείπουν πάνω από 50 90.000 οδηγοί και αυτή η έλλειψη πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της ευελιξίας και καλύτερων ε, συνθήκων εργασίας. Πολύ ωραία, το λόγο έχει ο κύριος Ερτούγκ για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο έθιξαν οι δύο προλαλήσαντες. Δηλαδή στο γεγονός ότι στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδρομους εντωμεταξύ έχουμε την εξής κατάσταση. Μάλλον μια κατάσταση που είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη και για τις χώρες που βρίσκονται οι αυτοκινητόδρομοι και για τις περιφέρειες αλλά και για εκείνους οι οποίοι καθημερινά δουλεύουν στους αυτοκινητόδρομους μακριά από την πατρίδα τους και μακριά από τις οικογένειές τους. Τούτο λοιπόν συμβάλλει σε αυτό που ήδη ελέγχθη, ότι αυτό το επάγγελμα δεν είναι πλέον ελκυστικό. Δεν πρόκειται μόνο για τα χρήματα τα χρήματα δεν είναι το μοναδικό διακύβευμα. Γιατί αν δει κανεί ε, τα έσοδα των οδηγών, κυρίω στην Νότια Ευρώπη, αυτά είναι πολύ ικανοποιητικά, πάνω από το μεσόρο. Αλλά και εκεί λείπουν οδηγοί. Άρα δηλαδή το διακύβευμα δεν είναι μόνο τα χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι συνθήκε είναι πολύ δυσάρεστες. Ξέρετε, αν βρίσκεται κανείς τρει μήνες καθοδόν, μετά ένα μήνα σπίτι του και μετά πάλι τρει μήνες καθοδόν, ε, κάποια στιγμή δεν θέλει κανείς ε, να ασκεί αυτό το επάγγελμα και γι' αυτό είναι σωστό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τη δέσμη μέτρων κινητικότητας υπαριθμών 1 και όπως πολύ σωστά επισήμαναν οι δύο συνάδελφοι προλαλήσαντες στον τομέα αυτό, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διαμορφωθεί ο τομέας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η κοινή αγορά να διατηρηθεί, να υπάρχει πρόσβαση στην κοινή αγορά, αλλά παράλληλα εκείνοι οι οποίοι μόνο μέσα από κοινωνικό ντάμπινγκ έφτιαξαν επιχειρήσεις, ε, αυτοί σε τελική ανάλυση να μην έχουν την απαραίτητη τη βάση, να τους την αφαιρέσουμε. Και υπάρχει η εξή κατάσταση. Πέρυσι, τον Ιούλιο, ψηφίσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο, απορρίφθηκαν και τα τρία θέματα που είχαν τεθεί για ψηφορία και μετά από ένα χρόνο ξανασχοληθήκαμε με τα θέματα αυτά. Ασχοληθήκαμε διακομματικά με τα θέματα αυτά και τελικά καταθέσαμε συμβαστικές προτάσεις. Βεβαίως, οι συμβαστικές προτάσεις δεν μπορούν να ικανοποιούν όλους. Ε, γι' αυτό λέγονται και συμβασμοί. Και γι' αυτό ήταν πολύ καλό το ότι επιτέλους μετά την 3η Δεκεμβρίου όταν προέκυψε στο Συμβούλιο ε, ομοφωνία, μάλλον έγκριση της, ε, των προτάσεων που είχαν κατατεθεί. Γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να καταθέσουμε αυτές τις προτάσεις και ε, αυτές οι προτάσεις ε, δυστυχώς ε, υπονομεύονται μέσα από τρίκ, πολλοί το προσπαθούν αυτό. Εκείνο όμως που παραμένει αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι χρειαζόμαστε αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Γιατί έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες οδηγών που περιμένουν αυτές τις ρυθμίσεις. Έχουμε σοβαρές επιχειρήσεις που, με, που συμπεριφέρονται πολύ σωστά στους εργαζόμενους τους και αυτές περιμένουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Αν λοιπόν αυτές δεν εγκριθούν, τότε θα συνεχιστεί η κατάσταση με τις γκρίζε ζώνες ε, θα εξακολουθήσει να υπάρχει διακατάσταση στους δρόμους και εντωμεταξύ θα υπάρχει και ο κίνδυνος ορισμένα κράτη-μέλη να λάβουν μονομερός μέτρα κάτι το οποίο θα ε, προκαλέσει την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γι' αυτό σας καλούμε να στηρίξετε τη συμβαστική μας πρόταση. Τι περιλαμβάνει η δική μου πρόταση. Εμείς προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα δύνατα σημεία της κείμενης νομοθεσίας, δηλαδή ε, μέσα σε τρεις μέρες ε, να μπορούν να γίνουν τρεις επιχειρήσεις, με συγγνώμη, 7 επιχειρήσεις. Αυτό όμως ε, ε, κρίναμε ότι δεν είναι σωστό, δεν μπορεί να ελεγχθεί και καταλήξαμε σε μια λύση που έγινε αποδεκτή και από τις ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Σε τελική ανάλυση είναι μια καλή προσέγγιση που νομίζω ότι της αξίζει και να υπερψηφιστεί. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων, ο κύριος Μπαχ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή Απασχόλησης που εργάστηκαν πάρα πολύ καλά και υπέβαλαν μια πολύ ωραία έκθεση. Δυστυχώς τώρα είναι σε ομοιρία η έκθεση για να ψηφιστεί όλο το πακέτο, όλοι οι δέσμοι. Δεν θα μπω στο περιεχόμενο. Οι συνάδελφοι Κιλόνεν, Βιν Βαντικάμ και Έρτουγκ έκαναν πολλά και σημαντικά. Θέλω να σκεγγραφίσω τώρα το θέμα όπως ε, βρίσκεται. Αν εγκαταλείψουμε το πακέτο θα δείξουμε ανευθυνότητα. Οι προϋποθέσεις ε, που περιγράφησαν ε, στους δρόμους δείχνουν ανευθυνότητα. Συνεχίζουν οι παράνομες και μη σοβαρές επιχειρήσεις. Καταστρατηγούν την ομοθεσία και, για να αποκομίσουν κέρδη. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ελπίζω την επόμενη εβδομάδα, αγαπητοί συνάδελφοι, να δείξουμε αίσθημα ευθύνης και να αποκαταστήσουμε την τάξη στους δρόμους μας με αξιοπρεπείς συνθήκες για τους οδηγούς. Και πάλι εκ μέρου τη επίτροπή ε, Απασχόληση και Κοινωνικών Θεμάτων, η κυρία Διαμπάλοβα, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, νιώθω προσωπικά μια μεγάλη απογοήτευση. Χάσαμε μια μοναδική ευκαιρία να θετήσουμε αποφάσεις ε, κέρια σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δυστυχώς δεν φάνηκε η υπευθυνότητα θα πρέπει να αλλάξουν κάποιοι κανόνε εν ώψη τη μεγάλη κινητικότητα στι μεταφορέ και χρειαζόμαστε του νέου κανόνε για να προστατεύσουμε του ε, οδηγού μα και τι επιχειρήσει ε, μεταφορών απέναντι στην αβεβαιότητα. Δεν θέλουμε κάθε χώρα να επιλέγει του δικού τη κανόνε και του δικού τη κανόνε εφαρμογή. Χάσαμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και κρίμα, συνάδελφοι. Και αντί να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει, κάνουμε ένα βήμα πίσω. Παλινδρομούμε. Ε, Έχουμε εσωτερική αγορά, μεταφορές, τα αγαθά που μετακινούνται από τα περνάνε τα σύνορα. Θα πρέπει να εφαρμόζονται σωστά ενιαίοι κανόνες. Ας αφήσουμε τη μικροπολιτική και ας επιστρέψουμε στην αναζήτηση συμβαστικής εφικτής λύσης. Θα έχουμε μια νέα ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό μας έχουν εκλέξει οι ψηφοφόροι μας. Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ο κύριος Βέλα. Μια στιγμή, μια στιγμή, συγγνώμη κύριε Βέλα. Κυρία Τλαπάγιοβα, υπάρχει μια ερώτηση με την μπλε κάρτα. Τη δέχεστε? Ωραία. Ο κύριο Κράμερ. Σήμερα είπατε το εξή, ότι τη Δευτέρα πήρατε 1620 τροπολογίε και είχατε δύο ώρε χρόνο για να αντιδράσετε, γιατί τότε θα είχε ε, εκπνεύσει η προθεσμία για άλλε τροπολογίε. Ξέρετε κάτι, τέτοια διαδικασία εγώ δεν την έχω ξαναδεί σε αυτό το κοινοβούλιο. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό μέχρι το μεδούλι. Βεβαίως ε, πρέπει να αναζητήσουμε συμβιβασμού, αλλά οι άλλοι σκιώδεις ηγητές ε, δεν συμφώνησαν και γι' αυτό είναι πολύ σωστό το ότι δεν θα αποφασίσουμε σήμερα. Εγώ δεν θέλω σε δύο ώρες να πρέπει να διαβάσω 1620 τροπολογίες και να κληθώ και να, αντιδράσω. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό και ε, δεν είναι αντάξιο ενός κοινοβουλίου. Κυρία Ντλαμπάγεβα, αγαπητέ συνάδελφοι, Πρώτα εγώ θα προτιμούσα μια ξεκάθαρη και σαφή ψηφοφορία. Αλλά τώρα είμαστε υπεύθυνοι. Έχουμε ευθύνε απέναντι στους οδηγούς και τις επιχειρήσεις μεταφοράς που αντιμετωπίζουν μια βεβαιότητα. Ακόμη και αν έπρεπε να ξοδέψουμε όλη τη μέρα και τη νύχτα στην προετοιμασία των τροπολογιών, θα πρέπει να το κάνουμε, να υπομιστούμε τι ευθύνε μα. Γι' αυτό μα εξέλεξαν. Ο κύριο Βέλα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη αξιότιμοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που ε, δεν ήμουν σήμερα παρόν. Βεβαίως η δέσμη μέτρων ε, κινητικότητας παραμένει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, κυρίως για την Επίτροπο Μπούλτς, αλλά δυστυχώς αναγκασμένη να συμμετέχει στο άτυπο Συμβούλιο Μεταφορών που λαμβάνει η χώρα στο Βουκουρέστι. Το Μάιο του 2017 2007 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρώτο τμήμα της δέσμης μέτρων κινητικότητας είχε ως στόχο κατά κύριο λόγο να βελτιωθούν οι συνθήκες στους δρόμους. Δεύτερον, να διασφαλιστεί ο θεμητός ανταγωνισμός, να αποφευθεί η κατάτμιση της κοινή αγοράς μέσα από ασυντόνιστους εθνικούς κανόνες και τρίτον, να περιστεί το διοικητικό άχθος ε, για τους άμεσα ενδιαφερόμενους, να υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι μέσω της ψηφιοποίησης. Έκτοτε λοιπόν έχει περάσει αρκετός καιρός, έχουμε προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, ε, κυρίως την κυρία Κιλόνεν, τον κύριο Βαντενκάπ και τον κύριο Ερτούγκ, οι οποίοι ήταν κινητήρες δυνάμεις σε αυτή τη διαδικασία. Ευθύς εξ αρχής γνωρίζαμε ότι αυτός θα ήταν μαραθώνιος, δεν θα ήταν σπριντάρισμα, δρόμος ε, ε, μικρής περιορισμένης, ε, περιορισμένων αποστάσεων. Γι' αυτό λοιπόν ήταν απαραίτητο να υπάρξει και μια ουσιαστική και ικανοποιητική περίοδος για να σκεφτούμε αυτούς τους κανόνες. Στο Συμβούλιο στις 3 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους Σκεφτήκαμε όλα αυτά και οι συγητές και οι σκιώδεις βρίσκονται πολύ κοντά σε μια καλή λύση στον τομέα των μεταφορών. Ο τομέας οδικός χρειάζεται μια ρηξικέλευτη λύση. Χρειάζονται μεταφορείς και η οδηγία ένα σταθερό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια. Αυτός ο τομέας δεν μπορεί να περιμένει περισσότερο. Μια συμφωνία στο Κοινοβούλιο, γρήγορη συμφωνία, θα καταδείξει ότι το Κοινοβούλιο θέλει να αντιμετωπίσει τα κατεπήγοντα προβλήματα του τομέα η εντατική εργασία του Κοινοβουλίου μας επέτρεψε να φτάσουμε σε μια λύση χωρίς ε, αμφισβητήσιμα σημεία, σημαντικές λύσεις, όπως οι εταιρείε εικονικές να καταπολεμηθούν, να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία με το εθνικών αρχών, καλύτερη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, όπως είναι ταχογράφη και ηλεκτρονικά έγγραφα φορτωτικές και κοινοποίηση και δήλωση από την πλευρά μεταφορέων και ε, επίσης κανόνες για ελαφρά οχήματα μεταφοράς. Αυτή η πρόοδο επέτρεψε στο Κοινοβούλιο να εστιαστεί στο τέλο στι συζητήσει στι τελευταίε εκκρεμότητε, δηλαδή κυρίω στους κανόνε περί καμποτά, ο χρόνο οδήγηση και ανάπαυση και τέλο εξίσου σημαντικό, πώ εφαρμόζονται οι κανόνε περί απόσπαση εργαζομένων στον τομέα δικών μεταφορών. Κατά την άποψή μα, οι συμβαστικέ προτάσει που υπευλήθησαν πετυχαίνουν σωστή ισορροπία και πετυχαίνουν του γενικού στόχου τη προτάσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλύτερε συνθήκε εργασία, καλύτερη επιβολή του νόμου, ε, λιγότερο διοικητικό άκτο για του μεταφορεί των εμπορευμάτων και χρήση τη ψηφιοποίηση. Σε αυτό το στάδιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, διατηρεί μια γενική επιφύλαξη, αλλά θα συνεχίσει να υποστηρίζει συζητήσει με σκοπό επίτευξη συμφωνία επ' αυτών των χαρτοφυλακίων προτεραιότητα. Μπορούμε να υποστηρίξουμε όλε τι τροπολογίε που διατηρούν την ισορροπία μεταξύ τη ελευθερία παροχή μεταφορικών υπηρεσιών βελτιώσεως των συνθήκων εργασίας και μείωση του διοικητικού άχθου από την άλλη. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω κάποιες σκέψεις σχετικά με συγκεκριμένα σημεία, ξεκινώντας από το λέξη Specialis όσον αφορά ε, την απόσπαση των εργαζομένων. Όταν η Γενική Οδηγία περί αποσπάσεως αναθεωρήθηκε, υπήρξε σαφής δέσμευση που ανελήφθη να θετηθούν ειδικοί κανόνες για τις οδικές μεταφορές το μοντέλο το ξεχωριστό για την απόσπαση ενώ ήταν διαφορετική από την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πετυχαίνει σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων των οδηγών από τη μια και την ελευθερία των εταιριών να παρέχουν διασυνοριακές μεταφορικές υπηρεσίες από την άλλη. Στηρίζεται από τον εισηγητή και περιέχεται στη γενική προσέγγιση που εθετήθηκε από το Συμβούλιο. Εν γέννη, υποστηρίζουμε τις απαιτήσεις περί για τον τομέα των οδικών μεταφορών, που είναι οι απλούστερες δυνατές συνθήκες που μπορούν να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Ε, φρονούμε ότι η προσέγγιση προωθήθηκε από την κυρία Κιλάνεν ε, πληρεί τους στόχους που ετέθησαν. Τώρα στρέφομαι προς τους κανόνες περιοδηγήσεως και αναπαύσεως και του χρόνου αναπαύσεως και οδήγησης είναι πολύ ευαίσθητο θέμα το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο όσον αφορά τι συνθήκε εργασία και την οδική ασφάλεια. Η άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ο οδηγό θα πρέπει να μπορεί ε, να έχει την εβδομαδία του ανάπαυση, μακρά ανάπαυση, είτε στο σπίτι του με την οικογένειά του ή σε άνετε συνθήκε, αλλά όχι στην, αίθουσα, καμπίνα οδήγηση. Θα πρέπει οι οδηγοί επίση να έχουν ασφαλή ε, δυνατότητα χώρου ανάπαυσης που είναι ασφαλή και αναπαυτική. Εξασφαλίζοντας έτσι η διαθεσιμότητα αυτών των χώρων ανάπαυσης είναι κάτι πολύ σημαντικό. Υποστηρίζουμε και ενεργούμε και προωθούμε ενεργά την ανάπτυξη ε, τομέων ε, περιοχών στάθμισης που είναι ασφαλή μέσω οικονομικής υποστήριξης από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας διαβεβαιώνω θετατικοποίηση της προσπάθειας που καταβάλει και μέσω χρηματοδοτήσεως τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μέσω του νέου μέσου για τη σύνθεση τη Ευρώπη. Για τη μεταφορά επιβατών, ο τομέα ε, πήρε μηνύματα σαφή τι τελευταίε εβδομάδε. Κανόνε περιοδηγήσεω και αναπαύσεω δεν είναι προσαρμοσμένοι όσον αφορά τη δραστηριότητα των οδηγών λεωφορείων και πούλμαν. Εισακούστηκε το μήνυμα που μα έστειλαν. Θα ξεκινήσουμε αμέσω μια πλήρη αξιολόγηση για ειδικού κανόνε για αυτού του οδηγού. Αν το ζητήσει το Κοινοβούλιο. Σίγουρα ο στόχος μας θα παραμείνει ο ίδιος. Βελτίωση συνθήκων εργασίας των οδηγών και η οδική ασφάλεια. Κλείνοντας, να αναφερθώ στους κανόνες για πρόσβαση στο επάγγελμα και στην αγορά. Όσον αφορά το καμποτάζ, είμαι ικανοποιημένο που η συγγήτρια διατηρεί την αρχή απεριόριστου αριθμού ε, επιχειρήσεων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κάτι που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καμποτάζ, ε, η περίοδος ε, ανάπαυση στο cooling, η περίοδος cooling off, όλα αυτά ήταν θέματα συζητήσεων ενδελεχών. Πρέπει να βρούμε σωστή ισορροπία. Η υποχρέωση τα φορτηγά να επιστρέφουν στο κράτος μέλος έδρας θα πρέπει να αξιολογηθεί μαζί με την, τα πρόσθετα κριτήρια εγκατάστασης και έδρας και τον νέο κανόνα απαιτεί οι οδηγοί να επιστρέφουν στο σπίτι τους τακτικά. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, προσβλέπω στη συζήτηση. Σας παρακαλώ να προβληματιστείτε προσεκτικά για πάνω στι σχέσεις των διαφόρων τομέων του πακέτου κινητικότητας. Απευθύνω έκκληση σε όλους να είναι επικοδομητικοί και να εστιαστούν επιλύσεων που μπορούν να εφαρμοστούν για τον τομέα οδικών μεταφορών και του εργαζομένου του τομέα και βεβαίω για την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ψηφοφορία θα είναι κρίσιμη για το έργο που μα περιμένει. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόπε Φοντανιά έχει τώρα το λόγο και μέρος τη Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω την θλίψη μου εδώ που δεν καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία μετά από τόσους μήνες δουλειά και γι' αυτό πρέπει να σας πω το πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποια είναι η πραγματικότητα που ισχύει στις μεταφορές, στις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά τις αποστάσεις που διανύονται και όσον αφορά και το χρόνο οδήγησης. Υπάρχει εδώ αντιπαράθεση μεταξύ χωρών σε βάρο του κοινού συμφέροντο του κλάδου. Φυσικά και είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε του εργαζόμενου και να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Όλοι το θέλουμε και γι' αυτό και προχωρήσαμε πολύ σε αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να γενικεύουμε και να χρησιμοποιούμε παράνομες πρακτικές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σαν άλοθη για τον προστατευτισμό τελικά. Η ελευθερία κυκλοφορίας ατόμων και εμπορευμάτων είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η προσφορά υπηρεσία επίσης είναι κάτι πολύ βασικό για την εσωτερική αγορά και για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε μια Ευρώπη με περισσότερη συνοχή τόσο στην επικράτεια όσο και οικονομική δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω και να βάζουμε φραγμούς στις ενδομεταφορές που ξοδέψαμε τόσο χρόνο για να τις καταργήσουμε. Ευχαριστούμε. Τώρα, εκ μέρους του ΕΛΚ, Ντέλη, για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, εδώ και δεκαετίες η εσωτερική αγορά και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών αποτέλεσε την ε, ηγετική δύναμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, μερικές χώρες έχουν εφαρμόσει εθνικά μέτρα τα οποία διχάζουν τελικά την ε, αγορά οδικών μεταφορών στην Ευρώπη. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν βοήθησαν να βελτιωθεί η κατάσταση. Αντίθετα, δίχασαν τις χώρες ακόμα περισσότερο ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Και είναι και πράγματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Εννέα χωρίς είναι κατά, υπήρχε μία αποχή στο Συμβούλιο, παρόλα αυτά προχώρησε η πρόταση. Τώρα ήρθε το πράγμα στο Κοινοβούλιο. Έχουμε τις αρχές, έχουμε τις αξίες, τις ευρωπαϊκές, αλλά συγχρόνως ένας από τους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών δηλαδή και η ενιαία αγορά, είναι πράγματα τα οποία τίθεται σε κίνδυνο εφόσον περάσει αυτή η πρόταση. Δεν είναι δυνατόν, αν δεν πετύχουμε σε οδικέ μεταφορέ, να έχουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά, γιατί θα είναι πιο ακριβέ οι μεταφορέ και τελικά θα είναι ο πολίτη αυτό ο οποίο θα πρέπει να πληρώσει. Πρέπει να ξαναβούμε σε διαπραγματεύσει, να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα πραγματικό σεβεβιασμό, κάτι το οποίο δεν έχουμε πετύχει τώρα. Είναι πολύ αργά, τελειώνει η θητεία μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολιτικέ ομάδε είναι διχασμένοι μεταξύ του. Δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε ήρεμα για αυτά τα θέματα πια. Έχουμε πάνω από χίλιε τροπολογίε. Μα ήταν δυνατό να καταλήξουμε σε λύση κάτω από αυτέ τι συνθήκε. Όχι, δεν το καταφέραμε για χρόνια τώρα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αναβληθεί αυτό το θέμα και να μείνει για την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλύτερα να μην έχουμε συμφωνία παρά να έχουμε μια κακή συμφωνία. Πρόεδρο, να τηρείτε το χρόνο σα, παρακαλώ, γιατί ο κατάλογο ομιλητών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, τώρα εκ μέρου των Σοσιαλιστών, για ένα λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι πολύ πραγματικά που δεν είναι εδώ η Επίτροπος Μπούλτσο. Νομίζω ότι έπρεπε να ήταν εδώ να μας ακούσει. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια στην έκθεση Κιλνόνεν και ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή δουλειά που καταφέραμε να κάνουμε με την εισηγήτρια και με τους υπόλοιπους συναδέρφους υπέρ της ενίσχυσης, γιατί αυτό είναι στη βάση της προσπάθειές μας, της ενίσχυσης των ε, ελέγχων φτάνουμε στην υποχρέωση του ταχογράφου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για το 2022 αλλά δεν θέλουμε να υπάρχουν διακρίσεις και να ενισχύεται η ξενοφοβία και ο προστατευτισμός. Δεν θέλουμε να φταίει ο οδηγός. Οι διάφορες δικήσεις θα πρέπει να διευκολύνουν τους ελέγχους, γιατί δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι φταίνει η οδηγή πάντα ε, και να είναι αυτή υπεύθυνη για τον έλεγχο ενό πακέτου εγγράφων. Είναι και επικίνδυνο στο κάτω-κάτω και δεν βοηθάει και στην αξιοπρέπεια του οδηγού. Τώρα το θέμα των ε, διεθνών μεταφορών και των αδομεταφορών. Εμείς είμαστε κατά του να επιστρέψουμε στην ε, αρχή, εκεί που ήμασταν ε, πριν. Χρειαζόμαστε βέβαια μια ευελιξία για τους οδηγούς αυτούς, τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους για παράδειγμα. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Ζήλε. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ταγιάννη χτες ε, το βράδυ για την αποφασή του, γιατί δεν είναι δυνατόν να νομοθετεί κανείς κάτω από αυτές ε, τις συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την περίπτωση θα φαίνεται σαν να είναι το... αυτός που ακολουθεί το Συμβούλιο σε αυτό που κάνει. Όχι, φυσικά και χρειάζονται συμβιβασμοί. Και το Κοινοβούλιο από τη στιγμή που δεν δέχτηκε το συμβιβασμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να πετύχει έναν υπεύθυνο και καλό συμβασμό. Και δεν πρόκειται μόνο για τώρα την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται για ολόκληρη αυτή τη θητεία. Πώς θα φαίνεται το Κοινοβούλιο με ένα τέτοιο πακέτο. Δεν είναι δυνατόν οι αρμόδιες επιτροπές να στέλνουν τέτοιες εκθέσεις όταν ακόμα και οι μεγάλες πολιτικές ομάδες δεν έχουν μια συγκεκριμένη θέση και όταν οι περισσότεροι θα κρατήσουν θέση αποχής. Αλλά ακόμα κι αν συνεχίζαμε τον επόμενο μήνα ε, δεν θα βοηθούσε και πολύ. Τι σημαίνει λοιπόν για τους πολίτες όλο αυτό παραμονή των ευρωεκλογών. Τι θα σκεφτούνε ότι θυσιάζουν την εσωτερική αγορά υπέρ των μεταφορών και υπέρ κάποιων εθνικών συμφερόντων για να επανεκλεγούν. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό θέλουμε να δείξουμε προ τα έξω. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα, ένα λεπτό. Για την Άντε. Ευχαριστώ. Η καλή λειτουργία των μεταφορών είναι κλειδί για την ανταγωνιστικότητα τη Ένωση. Αυτό το πακέτο κινητικότητα είναι θεμελιώδη στοιχείο για να αποφευθεί ο κατακαιρματισμό που προκαλείται από το εσωτερικό κοινωνικό ντάμπινγκ και από τις διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά για τους διαφόρους ε, που λειτουργούν στον ε, τομέα αυτό. Πρέπει να έχουμε κοινέ λύσεις λοιπόν, να μην υπάρχουν λύσεις από κράτος σε κράτος ε, που αυξάνουν τα προβλήματα. Γι' αυτό στηρίζω τις συμβαστικές προτάσεις που υπέβαλαν οι εισηγητές αυτών των τριών εκθέσεων. Αυτά που προτείνουμε βελτιώνουν την κατάσταση για τους οδηγούς, για τον κλάδο, βελτιώνουν την ασφάλεια των οδών, και προετοιμάζουν το μέλλον, ούτω ώστε σύντομα να έχουμε την ε, ψηφιοποίηση και την κατάργηση των οξυδίων του άνθρακα. Αλλάζουμε δηλαδή τη ζωή προς το καλύτερο. Γι' αυτό μας εκλέγουν ε, οι συμπολίτε μας. Αλλά ξέρετε ότι το καλύτερο είναι εχθρό του καλού. Αυτό ισχύει και στις μεταφορές. Γι' αυτό όσοι επιχειρούν να φρενάρουν για λόγου καθαρά εκλογικού, κάνουν λάθο. Δεν είναι φυσικά το βέλτιστο αυτό το πακέτο. Αλλά προβλέπει επαρκή συμφωνίες για να είναι πολύ καλύτερο από αυτά που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Και για δύο λεπτά τώρα για τους πράσινους η κυρία Αντέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και μήνες εργαζόμεθα για να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των ε, μισθωτών στις οδικές μεταφορές. Μήνες τώρα αυτοί οι μισθωτοί είναι θύματα ορισμένων ε, στο όνομα των συμφερόντων των χωρών τους. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες που εργάζονται με συνθήκες πολύ δύσκολες, ε, κουραστικές, δεν βλέπουν την οικογένειά τους, κοιμούνται σε πάρκινγκ, ε, τα αυτοκίνητά τους δεν συντηρούνται καλά, ορισμένοι κοιμούνται στα κουβούκλια των φορτηγών, υπάρχει οργανωμένο κοινωνικό ντάμπινγκ από τις μεγάλες εταιρείε του κλάδου που τους εκμεταλλεύεται μέχρι την πλήρη εξάντλησή του με τρομερές επιπτώσει για την οδική ασφάλεια. Ένας κουρασμένος οδηγό ε, στους δρόμους μας είναι κίνδυνος και για τον εαυτό του και για το φορτίο του αλλά και για όλους τους άλλους χρήστε. των οδών. Πρέπει να αρνηθούμε ω Κοινοβούλιο να εγκρίνουμε την εκμετάλλευση των εργαζομένων στον τομέα αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εδώ μέσα. Θα πρέπει να αρνηθούμε αυτά που είναι καθαρά μία σύγχρονη μορφή δουλείας στους αυτοκινητοδρόμους μας. Δεν υπάρχουν ε, ισότιμες συνθήκες εργασίας. Αυτό πρέπει να υπάρξει για όλους όσους εργάζονται στον κλάδο, στην Ένωση. Δεν θέλουμε ε, εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, ούτω ώστε η απόσπαση να ισχύει για όλους και όχι μόνο για ορισμένα επαγγέλματα. Δεν θέλουμε εξαντλημένους οδηγούς στους δρόμους μας γιατί έτσι κινδυνεύουμε όλοι, κινδυνεύει η ζωή μα. Γι' αυτό αρνούμεθα κάθε εξαίρεση από την απαγόρευση τη εβδομαδιαία ανάπαυση στο κουβούκλου. Δεν θέλουμε κοινωνική ζούγκλα. Δεν θέλουμε να γίνεται ό,τι να είναι. Ούτε αυτοκίνητα που επιστρέφουν άδεια στην έδρα του. Γι' αυτό θα αγωνιστούμε ούτω ώστε να εξακολουθήσει να ισχύει το καμποτάζ με βάση κανόνε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση <clears throat> πρέπει να τηρήσει τι υποσχέσει τη. Όλοι θέλουν μια κοινωνική Ευρώπη ε, ας την ε, επιδιώξουμε λοιπόν. Θέλουμε ο καθένας και το απαιτούμε να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του, όχι να ασχολείται με τα συμφέροντα τη χώρα του ή κάποιων χωρών. Είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε τι, τη σωστή εφαρμογή των ισχυών των κανόνων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Και τώρα για την ΚΟΕ η κυρία Γκονθάλεθ Πένιας. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είναι δυνατόν ότι οι σκληρές ε, ε, συνθήκες εργασίας να είναι πρόσχημα για να επιτρέψουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ, να επιτρέψουμε, να επιτρέψουμε διακρίσεις μεταξύ των οδηγών. Ορισμένοι συντηρητικοί λένε ότι αν θέλετε η εβδομαδιαία ανάπαυση να γίνεται με αξιοπρεπείς συνθήκες εκτός του οχήματο, τότε να πληρώνετε λιγότερο ένας Ισπανός οδηγός όταν οδηγεί εκτός Ισπανίας. Μα τι είδο εκβιασμού είναι αυτό. Θα πρέπει να υπάρξουν σωστοί κανόνε που να επιτρέπουν οι οδηγοί να μπορούν να κοιμηθούν σε ένα αξιοπρεπέ δωμάτιο όταν αναπαύονται. Να μην εργάζονται για πάνω από δύο εβδομάδε συνέχεια μακριά από τον τόπο προέλευσή του. Τα οχήματα να έχουν ε, ευφυεί ταχογράφου για να σταματήσουν οι απάτε και να μην υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό που σημαίνει ότι στέλνουμε οδηγούς στο εξωτερικό για να τους πληρώνουμε λιγότερο. Είναι θέμα αξιοπρέπειας, ισότητας ε, εργασιακών δικαιωμάτων και είναι και θέμα οδικής ασφάλειας. Ευχαριστώ. Νταμάτο, EFTD, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, η μεταφορά, το μέσο των μεταφορών χρειάζεται σημαντικέ απαντήσει κατεπηγόντω για να αντιμετωπιστούν τα διάφορα προβλήματα που είναι πολλαπλά. Καθημερινά βλέπουμε την πραγματική σκλαβιά που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε όλη την Ευρώπη. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να περνάνε τη ζωή του στα μεταφορικά μέσα, τρώγοντα, κοιμώντα εκεί, χωρί να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στο σπίτι του και να περάσουν τον χρόνο του με, με την οικογένειά του. Άλλο πρόβλημα του κοινωνικού ντάμπινγκ είναι ένα πρόβλημα του ανταγωνισμού, τα θέμη του. Θα πρέπει να επιτρέψουμε στι εταιρείε να μπορούν να ανταγωνιστούν ισότιμα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο τη ε, μεταγκατάσταση, να δώσουμε κινήτρα για ε, ισότιμα φορολόγηση και μισθολογικά. Ε, είδαμε τελευταία χρόνια μια τάση που μείωσε όλο και περισσότερο τα κοινωνικά πρότυπα, τα επίπεδα των μισθών. Τάση που σήμερα είναι απαραίτητο να επανεξισορροπηθεί. Είναι η δική μα ευθύνη σε αυτή τη θητεία, για αυτό το κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, θα πρέπει να δοκιμάσουμε το τέλο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Μεταφορών, να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν κανόνα, κοινωνικά, μια ρύθμιση και κοινωνικά δικαιώματα στου μεταφορεί μα στο μεταφορικό τομέα. Μάγερ για το ENF για ένα λεπτό. Ορίστε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, να μιλάτε ειλικρινά στους συμπολίτε μας. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να αποφασίσουμε ε, σωστά. Το πακέτο κινητικό το 1 δεν θα αποφασιστεί κατά την τρέχουσα θητεία. Δεν θα αποφασιστεί. Αυτό είναι λυπηρό βεβαίως για πολλού οδηγού σε όλη την Ευρώπη. Γιατί ποια είναι η κατάσταση τώρα λοιπόν. Δεν έχει υπάρξει μεγάλη αλλαγή από τότε που παρουσιάστηκε αυτό το πακέτο πριν από ένα χρόνο. Και τελικά τι επιτυχάνουμε. Το αντίθετο από αυτό που θέλαμε. Θέλαμε βελτίωση των συνθήκων εργασία των οδηγών. Η Αυστριακή Προεδρία υπέβαλε κάποιε προτάσει, ε, υπήρξε μια γενική προσέγγιση, αλλά δεν κατέληξε πουθενά. Και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, Υπάρχουν αντιδιαμετρικές, ε, αντιδιαμετρικές απόψεις μεταξύ ΕΛΚ και σοσιαλιστών. Αντιδιαμετρικά αντίθετες. Και από την άλλη μεριά, οι πράσινοι από την αρχή με χαοτικό τρόπο έχουν παρέμβει και με τρόπο που είναι αντιδημοκρατικός. Υπήρξαν και ανεπίσημες συνεδριάσεις των συντονιστών όπου δεν, έχουν, ε, είχαν, δεν είχαν προσκληθεί όλοι οι συντονιστές. Σας άκουσα κύριε Αντέλη Κύριε Μάγερ, δέχεστε μία μπλε κάρτα από την κυρία Ντέλη. Τι δέχεστε. Ωραία, παρακαλώ. Δεν δέχομαι σε αυτό το κοινοβούλιο να αμφισβητούμε τις ε, δεξιότητές μου και τις ικανότητές μου στην Επιτροπή Μεταφορών. Ε, λοιπόν, η ομάδα σας μάλιστα θέλει να ξεριζώσει Θέλει πραγματικά να επιδεινώσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και γι' αυτό στην Επιτροπή μου, στην προεδρο, θα κάνω τα πάντα για να βελτιώσω τι συνθήκε εργασίας των μισθωτών. Σα το λέω κοιτάζοντα κατάματα. Δεν ξέρω ποιο θεωρείτε ότι είστε για να κρίνετε εσεί την ποιότητα κυρίω τη Προεδρία μου. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν θα το δεχτώ. Φτάνει. Δεν ήταν ερώτηση. Ο κύριος Μάγερ έχει 30 δευτερόλεπτα να απαντήσει. Κυρία Αντέλη, θα πρέπει να δεχθείτε την κριτική. Ξέρετε ότι κάνατε ανεπίσπες συνεδράσεις συντονιστών χωρίς να καλέσετε όλους τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Γιατί μου λέτε και ποιος νομίζεις ότι είσαι. Εσείς ε, ποια είστε όταν ε, οργανώνετε οργανώνετε τέτοιες αντιδημοκρατικές και ανεδείς συναντήσεις. Κοιτάξτε, δεν έχουμε συζητήσει επί τη ουσία μέσω των καλαζίων καρτών. Η κυρία Λουκατσεύσκα λοιπόν έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να απευθύνω έκκληση προς την Πρόεδρο και όλες τις πολιτικές ομάδες. Ας μη χρονοτριβούμε πλέον ασχολούμενοι με αυτό το πακέτο κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Έχουμε πάνω από 1500 τροπολογίες. Είναι αδύνατο να πετύχουμε συμβιβασμό που έχει νόημα. Δεν είμαστε έτοιμοι να ετοιμάσουμε το πακέτο της κινητικότητας, ούτως ώστε να σαφές, αξιόπιστο, διαφανές και να σέβεται την ενιαία αγορά περιορίζοντας τον αθέμητο ανταγωνισμό. Επίσης δεν είμαστε σε θέση να φροντίσουμε ούτως ώστε το κόστος εφαρμογής να μην πλήξει τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Ε, συμφωνώ με την κυρία Ντελή, δεν θα πρέπει να εξετάζουμε μόνο τα συμφέροντα των χωρών μας. Νομίζω ότι μπορούμε να προσχωρήσουμε σε την πολιτική. Κυρίες και κύριοι, τι αυτό που συμβαίνει ε, είναι πονίδιστο αυτό που συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει τα διάφορα προβλήματα και τις ατασταλίες και τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν. Τι γίνεται όμως με τα κενά δρομολόγια, δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν τα δρομολόγια χωρίς φορτίο. Ε, και τι γίνεται με την απόσπαση των εργαζομένων στο μεταφορικό τομέα. Συμφωνήσαμε από αυτού και μετά θέλετε να περιορίσετε τον τομέα των μεταφορών και την επιστροφή στο χώρο διαμονής, στον τόπο διαμονής για πέντε ημέρες. Τι γίνεται με διαμονή σε ξενοδοχείο. Δεν έχουμε αυτά τα ξενοδοχεία και δεν έχουμε χώρου στάθμευση οι οποίοι να είναι ειδικοί για το σκοπό που θέλουμε. Και εγώ σα και όδης εισηγήτρια ήμουν έτοιμη να κάνω το στο... Κύριο Κασεύκα, Διακόπη ομιλήτρια. Κυρία Λουκασεύσκα, υπάρχει μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Ράτκα. Το δεχόσαστε. Δεχόσαστε την κάρτα. Ορίστε κυρία. Ναι. Δύο συγκεκριμένε ερωτήσει προ τη συνάδελφο. Πρώτον, όταν ε, αναφέρεστε ε, με τόσο παθιασμένο τρόπο στην ε, ελευθερία της εσωτερικής αγοράς τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι ελεύθερη από κοινωνικού κανόνε η εσωτερική αγορά. Και δεύτερον, όταν λέτε ότι επίκυνται οι εκλογέ, πόσο πρέπει να συζητάμε ένα τέτοιο νομοθέτημα πριν το θεωρήσουμε όριμο για να ε, ψηφιστεί. Γιατί ε, θα εκλεγούμε αν δεν θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας των οδηγών. Εγώ μίλησα με Ρουμάνους και Πολωνούς οδηγού σε γερμανικά και μου είπαν ότι οι συνθήκε του είναι άθλιε. Η κυρία Γιουκαζεύσκα, 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε, ε, προσπαθήσαμε μέσω τριμερών διαλόγων να το επιτύχουμε αυτό, αλλά για το καμποτάζ Όταν κάποιο δεν εργάζεται στη χώρα ε, προέλευσή του ή είναι απόσπαστο, όταν είναι κανεί μακριά από την ε, αιστεία του, γιατί θέλετε να το περιορίσουμε. Γιατί αυτή η διαμετακόμιση να θεωρείται απόσπαση. Ε, ένα αυτοκίνητο που εργάζεται με αυτόν τον τρόπο δεν εξυπηρετεί. Κύριε Ντεμόντε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να παρατηρήσω ότι πρέπει να αλλάξουμε το όνομα του πακέτου. Από πακέτο κινητικότητας πρέπει να το περάσουμε να το λέμε πακέτο ακινησίας. Εδώ και μήνες συνεχώς βλέπουμε να, να, να το μεταξύ Ολομέλειας και Επιτροπής Μεταφορών να πετάγεται το θέμα και θα πρέπει να ψηφίσουμε, αλλά αντί να ψηφίσουμε πρέπει να συζητήσουμε. Έγινε καλή δουλειά μέχρι τώρα νομίζω. Νομίζω ότι πετύχαμε κάποιες συμβαστικές λύσεις για το καμποτάζ, για την απόσπαση, για τους κανόνες περί χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης. Έχω κάποια προβλήματα όσον αφορά το διασυνοριακό καμποτάζ, διότι πιστεύω ότι επιτρέπει να υπάρξουν απάτες, αλλά συνολικά νομίζω ότι πραγματικά σημειώσαμε πρόοδο και θα πρέπει σίγουρα να φτάσουμε ε, στο να εφαρμοστεί ευφυής ταχογράφος, διότι μόνο έτσι ε, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε ακριβώς ότι τηρούνται οι προδιαγραφές. Απευθύνω έκκληση ε, μέχρι το τέλος της θητείας να ψηφιστούν αυτά, διότι μόνο έτσι θα μπορούμε να πούμε ότι εργαστήκαμε καλά για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Για 1,5 λεπτό, ο κύριος Σνοτόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, για τι πράγμα συζητάμε εδώ τώρα. Συζητάμε για τις συνθήκες εργασίας των οδηγών, ε, για τις συνθήκες ανάπαυσής τους, μιλάμε για τους ταχογράφους και ο Θεός ξέρει τι άλλο. Όμως όλοι αντιλαμβανόμαστε πάρα πολύ καλά ότι τελικά δεν πρόκειται για όλα αυτά τα θέματα στην ουσία. Γιατί οι οδηγοί φορτηγών διαμαρτύρονται μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Όλο αυτό το πακέτο κινητικότητα δεν είναι για καμιά βελτίωση προ όφελο των οδηγών. Για ένα και μόνο πράγμα πρόκειται. Πρόκειται για τι χώρε ε, τη περιφέρεια τη Ευρώπη, Ανατολική αλλά και Νότια Ευρώπη, για να ξεφύγουν από του κανόνε τη κοινή αγορά. Όλο αυτό το πακέτο κινητικότητα δεν είναι για τι συνθήκε εργασία, δεν είναι για τι συνθήκε οδήγηση. Είναι απλώ και μόνο για να διχάσει την κοινή αγορά, την εσωτερική αγορά. Κυρίες και κύριοι, οι χώρες που μπήκανε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκαν το γεγονός ότι υπήρχε μια εσωτερική αγορά και ανέπτυξαν τον κλάδο των μεταφορών τους και τώρα τους αποκόβουμε όλα αυτά τα θέματα δεν είναι αυτά που διακυδεύονται σήμερα. Να συζητήσουμε και αυτά, αν θέλετε, αλλά να καταλήξουμε και σε ένα συμβασμό. Τι συμβασμό είναι αυτό, αν υπάρχουν 600 τροπολογίε που πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα καλύτερο συμβασμό. Αυτό δεν είναι συμβασμό καθόλου. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να ψηφίσει σήμερα. Να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την επόμενη θητεία. Ευχαριστούμε. Υπάρχει μπλε κάρτα από τον κύριο Ερτούκ για σας. Κύριε Σλοτόφσκι, δέχεστε. Ευχαριστώ τον συνάδελφο. Συνάδελφε, θέτω το ερώτημα. Επειδή η συζήτηση μοιάζει να σημαίνει ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι πήραν το λόγο προηγουμένως ε, έλειπαν τους τελευταίους μήνες αλλά αυτοί ήταν ε, μαζί εδώ με του συναδέλφου Λουκασέφσκα, Τέλ, Ντέλη, Κίλονεν, μαζί συμφωνήσαμε τους συμβασμού. Τι είναι τώρα αυτές, ε, αυτά που λέτε, ήσασταν παρόντε. Στην αρχή ήταν υπέρ και μετά στραφήκατε κατά. Αυτή είναι η αλήθεια. Βλωτόφσκι. Απάντηση. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε αγαπητέ συναδελφοί, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε σήμερα. Ναι, είναι αλήθεια ότι εγώ στήριξα τους συμβιβασμούς και οι συμβιβασμοί αυτοί απορρίφθηκαν τελικά πέρυσι από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα δεν μιλάμε για συμβιβασμούς όμως καθόλου. Σήμερα μιλάμε για επίμαχα ε, ζητήματα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που οδηγούν στον διχασμό και την καταστροφή αυτής της εσωτερικής ε, αγοράς που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι για την απόφαση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί σε τι θα οδηγήσει την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε τις ίδιες τροπολογίες που θα επανακατατεθούν. Δεύτερον, λυπούμε που ο πρόεδρος δεν έκανε την προσπάθεια να απαντήσει σε επιστολή ε, διάφορων συναδέρφων και να είμαι δικιά μου, ερτού κτλ. Ε, όπου προτείνουμε ένα συγκεκριμένο σενάριο και συμβασμού. Ναι, έχουμε πάρα πολλέ τροπολογίε. Επίτηδε όμω έγινε αυτό. Να είμαστε ειλικρινεί, μην κορυδεύουμε του εαυτού μα. Επίτηδε κατατέθηκαν τόσο πολλέ τροπολογίε για να περιπλεχθεί η διαδικασία. Περί αυτού πρόκειται και πολλοί από εσά το επιβεβαιώσατε σήμερα γιατί λέτε να αναβληθεί. Ε, όχι. Έχουμε ε, συμβιβασμούς και την επόμενη εβδομάδα ε, θα ξέρουμε αν θέλουμε τελικά εσωτερική αγορά όπως προτείνουμε εμείς που να λειτουργεί που θα λύνει διάφορα ζητήματα, θα ενισχύει κοινωνικά δικαιώματα ή αυτό ή θα οδηγηθούμε σε μονομερή μέτρα, το οποίο είχαμε και κατά το παρελθόν και το οποίο οδηγούν σε κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς. Με δική σας ευθύνη. Ευχαριστούμε. Έχω δει ότι έχουν ζητήσει διάφοροι μπλε κάρτα. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Τέιλορ, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ένα μισή λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρό να ξαναδούμε τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Κάθε εργαζόμενο λέει η χάρτα αυτή, έχει δικαίωμα σε αξιοπρεπέ συνθήκε εργασίες που θα προστατεύουν την υγεία του και την αξιοπρέπειά του. Γνωρίζουμε όμως ότι στην περίπτωση μεταφορών ε, που διανύουν μεγάλες αποστάσεις, αυτές οι συνθήκες ούτε την υγεία προστατεύουν, ούτε την αξιοπρέπεια των οδηγών προστατεύουν, ούτε τίποτα. Πρόκειται για κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία τελικά καταπατούνται από εργοδότες. Πάρα πολλοί οδηγοί πρέπει να αναπαύονται στις καμπίνες τους χωρίς να έχουν πρόσβαση σε βασικά πράγματα, σε τουαλέτες ας πούμε. Οπότε το θέμα ε, δεν είναι απλώς δικαιώματα ή όχι, είναι και θέμα ασφάλειας, οδικής ασφάλειας. Γιατί αν δείτε τις στατιστικές βλέπετε ότι η κόπωση των οδηγών είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγεί σε ατυχήματα στον δρόμο. Οπότε το κόμμα μας η ομάδα μας θέλει να υπάρχει η περίοδος αναφοράς των δύο εβδομάδων και δεν ενθαρρύνουμε ε, αύξηση στο χρόνο οδήγησης. Και επίσης η μεγάλη διάρκεια ανάπαυση θα πρέπει να είναι σαν ένα ξενοδοχείο. δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ε, τροπολογίες. Δεν είναι υπεύθυνο, όπως είπανε και άλλοι συνάδελφοι. Διακόπτη πρόεδρος. Γιατί τελικά δεν καταλήξουμε σε τίποτα. Ευχαριστούμε. Είπα ότι δεν θα δεχτώ άλλε μπλε κάρτες επειδή έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ από σήμερα το πρωί. Ε, κυρία Κάρη, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, φέτος συναντήθηκα με οδηγούς από τις Φιλιππίνες. Μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλήσαμε για τις άδειε που δίνονται στους οδηγούς αυτούς και συζητήσαμε επίσης και για τους μισθούς τους, 15 δανέζικες κορώνες ε, την ώρα. Ε, καταλαβαίνετε ότι έχουν τελικά καλύτερες απολαβές, μπορούν να ζήσουν, μπορούν αξιοπρεπώς να ζήσουν με τα χρήματα αυτά. Και αναρωτιούνται αυτοί οι οδηγοί, γιατί οι δικοί μας. Γιατί έχουν τόσο κακές συνθήκες. Οι συζητήσεις αυτές έγιναν και ξανά έγιναν. Και έχει να κάνει και με τους δρόμους της Ευρώπης όπου κάπου 16 ώρες περνάνε στα φορτηγά τους οι οδηγοί οδηγότες και είναι φυσικά εξαντλημένοι στο τέλος. Αυτές είναι εμπειρίες που έχουμε. Μιλάμε για την εσωτερική αγορά εδώ στην Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση για το χρόνο οδήγηση. Θα το κάνουμε ή θα υποστηρίξουμε τι χώρε μέλη. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι μεταρρυθμίσει για το καποτάζ, η απόσπαση των οδηγών και ο χρόνο εργασία, αυτό το πακέτο δηλαδή κινητικότητα, ένα πράγμα δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο κοινωνική όσο ήταν οι δημοκρατικέ, οι σοσιαλιστικέ δημοκρατίε τη Ανατολική Ευρώπη. Πέρασαν 18 μήνε διαλόγου των κοφών. Και η νομοθετική κολλησιεργία των τελευταίων ωρών δείχνει για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να βελτιώσει τι συνθήκε εργασία των εργαζομένων τη. Και αποδεικνύει επίση ότι είναι τα οικονομικά συμφέροντα των χωρών που βρίσκονται σε ανταγωνισμό ένα με το άλλο ήθελε σώνει και καλά από ιδεολογία και από